Ξεκινάει η συνεδρίαση της Επιτροπής. Πρώτα δύο σημεία έχουμε να ψηφίσουμε όσον αφορά την απλουστευμένη διαδικασία όσον αφορά δύο θέματα. Οι παλιές ε, πράξεις στον οθετήμα του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική στην προηγούμενη συνεδρίαση στην Επιτροπή αποφασίσαμε, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί απλουστευμένη διαδικασία για το συγκεκριμένο τομέα σύμφωνα με αυτά που, ορίζει το άρθρο 45 παράγραφος 47 παράγραφος 1 αν πέντε μέλη συμφωνούν εγκρίνεται άνευ η ε, έκθεση έτσι είχαμε αποφασίσει συζήτηση, τώρα το χρησιμοποιούμε. Μιλάμε για τι επιτυχημένε πράξει του ε, Συμβουλίου στον τομέα τη κοινή αγροτική πολιτική. Υπάρχουν αντιρρήσει. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, η έκθεση υιοθετείται. Αναλόγως, δεύτερη ψηφοφορία αφορά την ανάθεση εργαστηριακών δοκιμών. Και εδώ στην προηγούμενη συνεδρίαση απλουστευτεί και να εφαρμοστεί η απλουστευμένη διαδικασία και αυτό το θέμα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που αναφέρει το άρθρο 46 παράγραφος 1, αν ένα δέκατο των μελών συμφωνεί, εγκρίνεται η έκθεση ανευτροπολογιών. Και εδώ σας ρωτώ αν υπάρχουν αντιρρήσεις. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, η έκθεση αυτή υιοθετείται. Και Πάμε στη διαδικασία του προπολογισμού που είναι στο σημείο 11, προπολογισμό 2010, τμήμα 3. Η συγγήτρια Ελίζαμπεθ Γέγκλ. Θα πρέπει να ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότηση όσον αφορά τον προπολογισμό 2010. Είχαμε ψηφίσει στην προηγούμενη συνεδρία τη Επιτροπή το τμήμα, το χρηματοδοτικό, το οικονομικό. Τώρα θα ψηφίσουμε τα κείμενα κατέφθασαν τροπολογίες όσον αφορά τις τροπολογίες πρέπει να ψηφίσουμε. Η κυρία Γέγκλ θέλει να πάρει το λόγο πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Κυρία Γέγκλ. Ναι. Όχι. Η κυρία Γέγκλ δεν θέλει να πάρει το λόγο και γι' αυτό ας ψηφίσουμε. Έχουμε τέσσερις τροπολογίες ε, για να ψηφίσουμε. Ξεκινάμε. Τροπολογία 1, παράγραφος 6α. Delange. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, Παπαστάμκου, του κ. Παπαστάμκου, παράγραφος 10. Υπέρ. Κατά, παρακαλώ. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Παπαστάμκος. Παράγραφος 10α. Υπέρ. κατά αποχές ναι. τελευταία τροπολογία κατά τμήματα πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος της τροπολογίας Λούλινγκ κατά αποχές πρώτο τμήμα εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα της τροπολογίας Λούλινγκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε και όλες τις... την τελική ψηφοφορία κάνουμε. Τελική ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ορότατα ομοφωνία. Σας ευχαριστώ. Οπότε... Αποχή Πόλσαν. Δεν έχουμε ομοφωνία δηλαδή. Υπάρχει μια αποχή. Η κυρία Γέγλε ζήτησε το λόγο. Έχετε το λόγο κυρία Γέγλε. Σας ευχαριστώ επιθυμώ να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους για την υποστήριξη που μου παρέσχουν για τις τροπολογίες του προϋπολογισμού. Επιθυμώ να ενημερώσω την Επιτροπή ότι έχουμε σε ό,τι αφορά τους αριθμούς ξεπεράσει το περιθώριο και σημειώνουμε και πάλι και εφόσον περάσουν στην ψηφοφορία θα έχει επιβεβαιωθεί Βεβαίω χρειάστηκε να κάνω κάποιες προσφορές ώστε να μπορέσει η Επιτροπή προπολογισμών να ξανακατέβει σε ορισμένα για να ξαναβρεθούμε μέσα στο περιθώριο. Μην απογοητευτείτε εάν εν τέλει στα νούμερα, στους αριθμούς δηλαδή που θα εγκρίνει η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα δείτε ότι ορισμένα κονδύλια έχουν ξανακατέβει. Είναι ωστόσο σημαντικά αυτά που επιτύχαμε και για τους γαλακτοπαραγωγούς. Σας ευχαριστώ κυρία Γέγκελ, ευχαριστώ όλους. Εάν συμφωνείτε, πάμε στο σημείο 12. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε τη χαρά να έχουμε την κυρία Λόριτς Χόφμαν, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Γενικής Διευθύνσεως Γεωργίας, η οποία θα μας κάνει μια παρουσίαση, γενική παρουσίαση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Πιστεύω, μεταξύ άλλων, θα ήταν χρήσιμο να σχολιαστούν οι εφαρμοστικές διατάξεις του καθεστώτος υγείας, της ε, ελέγχου υγείας της κοινή γεωργική πολιτική και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την ανάκαμψη τη οικονομία στα πλαίσια πολιτική ερωτική ανάπτυξη. Η κυρία Λόρι Χόφμαν θα έχει το λόγο πρώτα και μετά θα ξεκινήσει μια συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχά να πω ότι η μονάδα για την οποία εργάζομαι ασχολείται με τις οριζόντιες πτυχές της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Αναλύουμε επίσης και προτείνουμε μελλοντικές πολιτικές. Ασχολούμαστε περισσότερα όμως περισσότερο με τις οριζόντιες πτυχές Υπάρχουν και οκτώ γεωγραφικές μονάδες που ασχολούνται συγκεκριμένα προγράμματα των κρατών μελών και επεξεργάζονται τα θέμα λεπτομερώς με τα κράτη-μέλη, επεξεργάζονται τα προγράμματα και πώς εκτελείται και υλοποιείται η πολιτική. Τώρα πάμε πίσω. Η πολιτική αγροτική ανάπτυξη ε, ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 τότε. Είχαμε κάποια μέτρα όπως υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών και είχαμε υποστήριξη για την ε, πρώιμη συνταξιοδότηση, υποστήριξη των νέων γεωργών. Τότε εξελίχθηκαν τα πράγματα, προσθέσαμε και άλλα μέτρα στις βασικές παρεμβάσεις, διότι υπήρχαν απαιτήσει προσαρμογής ε, για τον τομέα της γεωργίας και απαιτήσει αυξανόταν, δηλαδή για αναδιάρθρωση ή στις αγορές. Ε, σήμερα ποια είναι η κατάσταση αλλάξαμε την προσέγγιση αρκετά όσον αφορά την περίοδο 2007 με 2013, αυτή που διανύουμε τώρα, και όσον αφορά αυτά που είχαμε πριν το 2007, είχαμε τρία ταμεία διαφορετικά που παρενέβαιναν στη, στα μέτρα αναπτύξεως της υπαίθρου, το Ταμείο Προσανατολισμού, του ΦΕΟΓΑ και τα διάφορα μέσα, τα οικονομικά για τα νέα κράτη-μέλη και εκεί συνδυάσαμε πέντε δυνατότητες προγραμματισμού στις περιοχές στόχου 1 έμπαινε η πολιτική του στόχου 1 στις περιοχές στόχου 2 πολιτικές του στόχου 2 και ξεχωριστό προγραμματισμό για άλλε περιοχέ ήταν μεγάλο βάρο για τα κράτη-μέλη. Υπήρχαν πολλά διαφορετικά συστήματα προγραμματισμού και διαχειρίσεω των προγραμμάτων, διαφορετικά οικονομικά συστήματα και διαφορετικούς κανόνες όσον αφορά τους ελέγχους και η υλοποίηση των μέτρων για να διευκολυνθούν τα πράγματα διότι τα κράτη-μέλη μας είπαν ότι είναι πολύ μεγάλο το άχθος για τη νέα περίοδο Βλέπετε στο κάτω μας εικόνα στη γίνεται έχουμε ένα, κάτι σαν κτίριο. Έχουμε ένα ταμείο που είναι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Ανάπτυξη Πέθρου και εκεί εντάσσονται όλα τα μέτρα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Και έτσι έχουμε έναν προγραμματισμό, σύστημα προγραμματισμού, ένα σύστημα υλοποίησεως, ένα διαχειρίσεως και ελέγχου. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη διότι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, το τρόπος διευκολύθηκε το έργο των κρατών μελών. Λοιπόν, τα ταμεία από τα οποία ξεκινάμε. Δεύτερο επίπεδο της εικόνας. Βλέπετε τους βασικούς στόχους της πολιτικής. Αντικατοπτίζονται στους άξονες στόχους, προτεραιότητες, μπορείτε να τους πείτε και έτσι. Πρώτα απ' όλα θέλουμε ανταγωνιστικότητα, αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Είναι σημαντική η ανταγωνιστικότητα για την γεωργία, για να προσαρμόστε η γεωργία στις διάφορες καταστάσεις, να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσει για προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς και επίσης να γίνεται καινοτόμα παραγωγή, να ακολουθούνται καινοτόμε προσεγγίσεις και σε κάθε άξονα προσφέρουμε διάφορα μέτρα μπορούν να διαλέξουν τα κράτη-μέλη για τα προγράμματά τους. Θα τα αναλύσω εκτενέστερα αργότερα. Έχουμε λοιπόν τον άξονα της ανταγωνιστικότητας. Στηρίζεται με μέτρα όπως εξυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων. Μπορούμε να υποστηρίξουμε δραστηριότητε για στην αγορά και μεταποιήσεως, αναπτύξεως νέων προϊόντων, νέων τεχνικών παραγωγής και συνεργασίας των διαφόρων εταίρων ούτως ώστε να καταλήξουμε σε νέα προϊόντα και νέες τεχνικές και παρέχουμε υποστήριξη για βοήθεια για φυσικές καταστροφές και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, κατάρτιση των ε, γεωργών. Τα τελευταία χρόνια φωτίστηκε ιδιαίτερα αυτό το θέμα και τονίστηκε. Διότι είναι ξεκάθαρο ότι πολλά μέτρα οργανώνονται καλά και υλοποιούνται σωστά και αποτελεσματικά μόνο αν οι γεωργοί ξέρουν πώς και τι να κάνουν. Άξον 2. Δεύτερος στόχος. Περιβάλλον και διαχείριση ε, της υπαίθρου. Εκεί Υπάρχουν ε, γνωστά μέτρα της αναπτύξεως της υπαίθρου, υποστήριξη των λιγότερο ευνοϊκών περιοχών, των περιοχών που είναι σε δυσχερέστερη θέση και εκεί πρέπει να αντισταθμίσουμε το υψηλότερο κόστος που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί, διότι είναι σε περιοχές, ασκούνται επάγγελμά του σε περιοχές ε, που εκτίθονται σε φυσικά προβλήματα λόγω περιοχής. Οι πληρωμές αντιστάθμισης των ορεινών περιοχών που είναι υποκατηγορία του τομέα αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντικές στις πληρωμές. Μετά υπάρχει δυνατότητα να υποστηριχθούν οι γεωργοί στα πλαίσια του Natura 2000. Εντάσσονται κάποιες αστεριότητες στη Natura 2000. Εκεί καταβάλλονται αποζημιώσεις σύμφωνα με συγκεκριμένε απαιτήσει ε, που πρέπει, προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για αυτέ τι περιοχέ, Κάποια μέτρα για τα δάση επίση προβλέπονται και τα σημαντικότερα μέτρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου είναι η αγροπεριβαλλοντική πολιτική όπου περίπου 20% του συνολικού προπολογισμού πάει εκεί. Μετά έχουμε και τον άλλο άξονα διασύνδεση γεωργίας με άλλους τομείς οικονομίας της υπαίθρου. Στόχος εδώ είναι να επιτρέψουμε στον αγροτικό τομέα να μπορεί να κινείται τρόπο και να συνδέεται και με άλλου τομεί, με άλλε Όπως ξέρετε, κάτι που προβλέπεται στον άξονα 2 είναι τουρισμός. Υπάρχει διασύνδεση μεταξύ Πέθρου και Γεωργίας. Η υποστήριξη υποδομών επίσης παρέχεται βασική υποδομή. Εδώ έχουμε τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, ευρυζωνικές υποδομές και άλλες δραστηριότητε ανακαίνιση χωριών, υποστήριξη μικροεπιχειρήσεων σε τομείς εκτός γεωργίας. Λοιπόν, έχουμε διάφορους στόχους. Και είναι ισορροπημένοι μέσα σε ένα πρόγραμμα οι τομεί. Γι' αυτό η νομοθεσία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να δαπανούν κάποιους πόρους στους τρεις τομείς. Τα κράτη-μέλη πρέπει να δώσουν 10% τουλάχιστον του κονδυλίου του ΦΕΟΓΚΑ για ανταγωνιστικότητα, 25% για περιβάλλον και διαχείριση των γεών και 10% για ποικιλομορφία και ποιότητα διαβίωσης. Όλα αυτά είναι στο leader που είναι ένας τρόπος εφαρμογής της πολιτικής. Δεν θα σε λεπτομέρειες. Βασίζεται σε τοπικές ομάδες δράσης που εφαρμόζουν σε τοπικό επίπεδο την αναπτυξιακή πολιτική, προσπαθούν να προωθήσουν την περιοχή τους. Αυτές οι ομάδες είναι κομμάτι του περιβάλλοντος, του τοπικού και παίρνουν αποφάσεις σχετικά με το πώς θα έπρεπε να αναπτυχθεί η περιοχή. Εμείς τους υποστηρίζουμε. Μπορούν να εφαρμόσουν αυτές οι ομάδες leader μπορούν να εφαρμόσουν πολιτικές των τριών αξώνων. Μπορούν να διαλέξουν τα μέτρα που θέλουν αλλά εστιάζονται, κατανοητό αυτό, κυρίως στον άξονα 3 σε αυτή τη φάση. Διότι αυτά τα μέτρα ε, βολεύουν πιο πολύ τη στρατηγική τους. Όλα αυτά υλοποιούνται μέσω μέτρων. Αναφέρονται στους άξονες. Βλέπετε τη διαφάνεια. Σχηματίστε μία εικόνα τώρα πώς θέλουμε να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτέλεσμα. Πώς μπορούν να εστιάσουν τις πολιτικές τους στα κράτη-μέλη για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες. Αν θέλετε θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον, είναι θέμα διατήρησης του τοπίου, αν θέλετε, βελτίωση της ποιότητας του χώματος, των εδαφών, ποιότητα, ποσότητα υδάτων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλα αυτά. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς όλα αυτά τα μέτρα που στρέφονται γύρω από αυτό το ελλειψοειδές στο κέντρο. Τα μέτρα προέρχονται από διάφορους τομείς, όπως βλέπετε, από διάφορους άξονες και εξυπηρετούν διαφορετικούς ε, στόχους. Μπορεί να έχετε κατάρτιση σε συγκεκριμένες επενδύσεις για εκμεταλλεύσεις για να έχει θετικά αποτελέσματα. Τα περισσότερα μέτρα προέρχονται από τον άξονα 2, από το πράσινο κομμάτι. Έχετε και άξονα 3, ανοιχτό γαλάζιο, μέτρα που εξυπηρετούν στόχους σχετικούς. Και μετά έχουμε την πολλαπλή συμμόρφωση από τον πρώτο πυλώνα, κάτι που λαμβάνεται υπόψη, που θεωρείται υποχρέωσης ετέλο, περαιτέρω πληρωμές. Τα κράτη-μέλη τι πρέπει να κάνουν για να εφαρμόζουν επιτόπου μέτρα. Για τη νέα περίοδο 2007-2013 θεωρήσαμε ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε μία προσέγγιση πιο στρατηγική. Διότι κατά το παρελθόν τι είδαμε. Ότι είχαμε πολλαπλά μέτρα. Έχουμε περίπου 40 μέτρα για την ανάπτυξη πέθρου. Και τα κράτη-μέλη επέλεγαν τα μέτρα διαδοχικά, το ένα μετά το άλλο. Ή χρησιμοποιούσαν πάντα τα ίδια μέτρα, έχοντας το λόγο τους βέβαια. Θεωρήσαμε ότι χρειάζεται στατηγικός προβληματισμός και αντιμετώπιση. Γι' αυτό, μαζί με τα κράτη-μέλη, αποφασίσαμε επί προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τη συγκεκριμένη περίοδο. Καθορίζουμε προτεραιότητες για την πολιτική αναπτύξεως αγροτική αναπτύξεω σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και αυτέ οι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω απορρέουν από τι γενικέ προτεραιότητε που έχουμε όσον αφορά τη βιωσιμότητα, αλλά όσον αφορά και τους στόχους ανάπτυξης και απασχόλησης της Λισαβόνας. Άρα τις διάφορες πτυχές τις μεταφέρουμε στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και τα κράτη-μέλη προέβησαν σε ανάλυση της υπαίθρου τους, ποιες ανάγκες υπήρχαν για προσαρμογή, τι έπρεπε να αλλάξουν και τα κράτη-μέλη ετοίμασαν εθνικά στρατηγικά σχέδια. Εκεί συμπεριλαμβάνουν αυτά που χρειάζονται τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και προσαρμόζουν τις προτεραιότητες αυτές στις ανάγκες κάθε κράτους μέλους. Έχω μια στρατηγική για κράτος μέλος, όπου το κράτος μέλος λέει πού πρέπει να εστιαστούν οι προσπάθειες στην επόμενη αυτή περίοδο. Και βάσει της εθνική στρατηγική, τα κράτη-μέλη προγραμματίζουν και αποφασίζουν ποια μέτρα διαλέγουν. Ποια είναι τα δεδειγμένα μέτρα, με άλλα λόγια, για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής τους. Μετά την έγκριση των προγραμμάτων, τα κράτη-μέλη εκτελούν και υλοποιούν Έχουμε επιτροπές ελέγχου, παρακολούθησης, αξιολόγησης. Γίνεται συνεχώς αξιολόγηση. Θέλουμε να δούμε σε ποιο βαθμό εκτελέστηκαν οι πολιτικές, αν χρειάζονται αλλαγές. Από αυτή τη διαδικασία είδαμε ότι έχουμε 27 εθνικές στρατηγικές εθνικά στατηγικά σχέδια, ένα για κάθε κράτες μέλος, αλλά σε επίπεδο προγραμματισμού Έχουμε κράτη-μέλη που επιλέγουν συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο και άλλα κράτη-μέλη που έχουν περιφερειακά προγράμματα. Για ομοσπονδιακές χώρες, Ισπανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί έχουν περιφερειακό πρόγραμμα, περιφερειακά προγράμματα και η Γαλλία έχει περιφερειακά προγράμματα. Οπότε φτάνουμε στα 88 προγράμματα εθνικά και περιφερειακά. Και έχουμε δύο εθνικά προγράμματα πλαίσια, Ισπανία, Γερμανία, που είναι γενικά πλαίσια για να κινηθούν τα περιφερειακά προγράμματα. Και έχουμε τέσσερα προγράμματα για εθνικά δίκτυα αγροτικής ανάπτυξης, διότι αποφασίσαμε ότι χρειάζεται ισχυρή δικτύωση, ούτως ώστε να γίνεται ανταλλαγή εμπειριών, ανταλλαγή απόψεων επί των πολιτικών. να υπάρχουν επαφές μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Έτσι, τα καλά παραδείγματα ανταλλάσσονται και οι δυσκολίες ανταλλάσσονται και συζητώνται. Έχουμε Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να έχουν και εθνικά δίκτυα δεν χρειάζεται όμως να τα διοργανώνουν πάντα στη μορφή που προβλέπουν τα προγράμματα. Γι' αυτό έχουμε μόνο τέσσερα προγράμματα. Τώρα για, τα... για τον προπολογισμό. 91 δισεκατομμύρια πάνω κάτω διετέθησαν για τα 27 κράτη-μέλη για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για αυτό το σκοπό εθνική συγχρηματοδότηση και εθνική συμπλήρωση ποσών, κρατικέ ενισχύσει, προβλέπονται σε κάποιες τομείς και έχουμε και ιδιωτικές δαπάνες, διότι για κάποια προγράμματα χρειάζονται και ιδιωτικά κονδύλια και κρατικά κονδύλια και τα κρατικά κονδύλια χωρίζονται σε αυτά που δίνονται σε κοινοτικό επίπεδο και σε αυτά που χορηγούνται σε εθνικό. Βλέποντα το συνολικό όγκο, στο συνολικό ποσό, πάμε στα 225 δις ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ γίνεται και διαφορά μεταξύ πολιτικής συγχρηματοδότησης και μη συγχρηματοδότησης. Υπάρχουν συνέπειες βέβαια, αλλά βλέπετε τι γίνεται. Έχουμε ένα αρχικό ποσό που συνοδεύεται από άλλους οικονομικούς πόρους και υπάρχει σημαντικό αποτέλεσμα, ε, σημαντικό φαινόμενο μοχλού, πολλαπλασιασμού δηλαδή των αποτελεσμάτων από αυτό το σύστημα. Εδώ βλέπετε πώς οργάνωσαν τη χρηματοδότηση τα κράτη-μέλη. Πώς διέθεσαν χρήματα για τους διάφορους στόχους, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Μεγάλα κομμάτια, άξον ένας, ένα συγγνώμη, είναι ανταγωνιστικότητα, αναδιάρθρωση, ενοτομία και περιβάλλον και το οποίο πάνω από 70%, 78% των πόρων πάνω εκεί. Και μετά έχουμε τον άλλο άξονα, τους άλλους άξονες με μικρότερα ποσά. Διαφέρει η κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη. Διαλέγουν οι χώρες τα μοντέλα τους. Άλλες κινούνται στην κατεύθυνση του άξονα 1, λιγότερο στον άξονα 2. Όλα εξαρτώνται από τις ανάγκες των κρατών μελών. Τώρα για το ναι, έλεγχο υγείας της αγροτικής πολιτικής, διεξήχθη αυτός και είδαμε ότι χρειάζεται προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Αλλάζει το περιβάλλον, αλλάζει η κατάσταση. Άρα χρειάζεται προσαρμογή. Επενδύσεις, μέτρα και άλλες δραστηριότητε στην Ήπεθρο. Και γι' αυτό Έχουν καθοριστεί προτεραιότητες. Πέντε βασικά σημεία. Και γι' αυτό για τι προτεραιότητε πρέπει να διατεθούν και άλλοι πόροι. Και υπάρχει μηχανισμός διαμόρφωσης που μεταφέρει χρήματα από τον πρώτο στο δεύτερο πύλωνα. Και ενισχύθηκε αυτός ο μηχανισμός. Είχαμε πριν αυτή την, ε, το μηχανισμό διαμόρφωση και κατανομής, ενισχύθηκε. 3,36 δις ευρώ επιπλέον διετέθησαν για προγράμματα αναπτύξεως της Γεωργίας για αλλαγή του κλίματος, διαχείριση των υδάτων, διεκπικυλομορφία, αναδιάθρωση που μπήκε λίγο αργότερα σε αυτό το τομέα. Δεν ήταν στην αρχική πρόταση. Και να πω ότι η προτεραιότητα ιδιαίτερη έχει καινοτομία, καινοτόμε πτυχέ που συνδέονται με τι διάφορε βασικέ προτεραιότητε. Το πακέτο ανάκαμψη το αποφάσισαν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ήθελαν κατεπίγουσα δράση, άμεση δράση. Μέχρι το τέλο του παρελθόντο έτου για να η οικονομική κρίση. Ούτω ώστε να γίνουν δημόσιε επενδύσει σε υποδομέ και άλλου τομεί, κυρίω τι υποδομέ όμω και περίπου άλλο ένα δις διετέθη για την, για την αγροτική ανάπτυξη. Για να βελτιωθούν οι ευρυζωνικές υποδομές στην Ήπεθρο. Διότι θεωρήθηκε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα αυτό. Το είδαμε από τα στοιχεία. Είδαμε ότι η Ήπεθρος εξυπηρετείται άσχημα στην συγκρίση με τις αστικές περιοχές όσον αφορά τις ευρυζωνικές υποδομές και εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι αυτό είναι σοβαρό μειονέκτημα για την Ήπεθρο. Και η βελτίωση της καταστάσεως θα επέτρεπε στην Ήπεθρο να καλύψει το κενό και να μπορέσει να αντισταθμίσει τις δυσκολίες και ανεπάρκειες που αντιμετωπίζει λόγω της ε, χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, την πούμε οικονομική κρίση στις διαπραγματεύσεις τελικά δημιουργήθηκε ένα άνοιγμα και το ένα δις ευρώ δεν είναι κάτι υποχρεωτικό. Δεν μπαίνει υποχρεωτικά για βριζονικές υποδομές. Μπορούν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα και για τις προαναφερθήσεις προτεραιότητες που εντοπίστηκαν στον έλεγχο υγείας της ΚΑΠ. Ποια είναι η κατάσταση τώρα. Μέσα Ιουλίου λάβαμε τις αλλαγές προγραμμάτων και περιφερειών που προβλέψαν τα κράτη-μέλη, διότι έπρεπε να πάρουν και άλλα ποσά από τη διαμόρφωση από το πρόγραμμα ανάκαμψη και να εντάξουν τα χρήματα αυτά στο πρόγραμμά του και τα χρήματα αυτά πρέπει να τα δώσουν για τι προτεραιότητε που εντοπίστηκαν. Έχουμε 88 προγράμματα που έχουν ενταχθεί και συνδυάσαμε τη διαδικασία ελέγχου της υγείας με τη ε, διαδικασία ανάκαμψης. Οπότε η αναθεώρηση πρέπει να γίνει πλευράς κρατών μελών άπαξ. Τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους, αλλά έχουμε πολλές πιέσεις και τα κράτη-μέλη πιέζονται. Το κουβεντιάσαμε σε διάφορες επιτροπές με τα κρατη το ξέρουμε. Και προσπαθούμε να εγκρίνουμε μέχρι το τέλος του χρόνου τα προγράμματα. Πρέπει. Έχουμε προϋπολογισμό κονδύλια για το 2009 που θα πρέπει να δεσμευτούν φέτος, να διατεθούν, διότι αλλιώς θα χαθούν. Είναι τα χρήματα από το πρόγραμμα ανάκαμψης, από το πακέτο ανάκαμψης. Υπάρχει ένα ποσό για το 2009, άλλο ποσό για το 2010. Το ποσό για το 2009 είναι 600 εκατομμύρια πρέπει να ενταχθούν στα προγράμματα και θα πρέπει να εγκρίνουμε και όλες τις αλλαγές ώστε να μπορέσουμε αυτά τα χρήματα να τα συμπεριλάβουμε στα προγράμματα. Τέλος, να σας δώσω μία εικόνα όσον αφορά το τι κάνουν τα κράτη-μέλη με τα χρήματα που παίρνουν από το πρόγραμμα, το πακέτο ανάκαμψης και από τον έλεγχο υγείας. Αυτή είναι μία αρχική εικόνα, διότι ακόμα συζητάμε με τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να δούμε αν είναι σωστή η λύση αυτή που ακολουθούμε. Αν οι, οι ανάγκες που αναφέρουν στρατηγικές είναι σωστές, αν καλύπτονται σωστά από τα προγράμματα και η εντύπωσή μας είναι ότι πάνω από ένα τρίτο των χρημάτων πηγαίνουν στη βιοπικιλότητα, σε αυτή την προτεραιότητα, μετά το 23% πάει στη διαχείριση των υδάτων, 15% για τα γαλακτοκομικά, μεγάλη μέρημνα των κρατών μελών αυτή, και μικρότερα ποσά πάνε σε άλλα θέματα, σε άλλε προτεραιότητε. 10% για ευρυζωνικέ υποδομές και για αλλαγή του κλίματος. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 6%. Αυτή είναι μια αρχική εικόνα. Βλέπετε τις επιλογές των κρατών μελών σε αυτή τη φάση. Αναφέρθηκα σε διάφορα θέματα εκτενώς, συγγνώμη, αλλά δεν θα μπορούσα να είμαι συντομότερη, θα ήταν πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Άριστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Χόφμαν, την ευχαριστούμε. Θερμό χαιρετισμό υποδοχής στην, ε, στα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας ε, του Κοινοβουλίου της ε, Βόρειας Ιρλανδίας. Ξεκινάμε τις ε, συζητήσεις της Επιτροπής. Ήδη ζήτησαν το λόγο. Ε, ε, ο κύριος Νίκολσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Απευθύνω και εγώ χαιρετισμό σε πρόσωπα από την εκλογική μου περιφέρεια στην Βόρεια Ελλανδία. Είναι κάπως τριμωγμένα βέβαια εδώ και οι συνάδελφοί μου κάθισαν εδώ και μάλιστα και χωρίς μετάφραση αλλά τουλάχιστον μπορούμε να μιλάμε τη μητρική μας γλώσσα. Καλώς ήρθατε λοιπόν εσείς φίλοι από τη Βόρεια Ιρλανδία. Τώρα, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και όλους όσοι συνεργάστηκαν για την παρουσίαση, που ε, τη βρήκα εξαιρετικά χρήσιμη για το ειδικότερο αυτό θέμα, που είναι ωστόσο σημαντικό. υποστήριξη δηλαδή για τις ε, αγροτικές περιφέρειες της υπαίθρου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί αγρότες βρίσκονται σε δύσκολη θέση και ε, αρχίζει και γίνεται αντιληπτό αυτό. Τώρα, από τότε που ε, εφευρέθηκε ο τρίτος πυλώνας και που τον προώθησε ο τότε Επίτροπος Φίσλερ, είναι, το πρόβλημα είναι ότι ποτέ δεν έδωσαν αρκετά χρήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεύτερο πυλώνα, συγγνώμη. Δεύτερο πυλώνα δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την αγροτική οικονομία, αλλά ποτέ δεν πρικοδοτήθηκε με επαρκή κονδύλια. Και ακόμα τώρα προσπαθούμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση και ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει. Διότι όλα αυτά τα χρήματα που είδατε στι οθόνε σήμερα είναι πολύ ωραία. Θαυμάσια να μιλάτε για ένα δισεκατομμύριο, αλλά γνωρίζετε κι εσεί καλά και βλέπω ότι νεύετε καταφατικά ότι κατανέμονται σε 27 χώρες μέλη, στις διάφορες περιφέρειες. Και μέχρι να φτάσει το κονδύλι ε, στον τελευταίο απολύπτη, το ποσό που έχει μείνει είναι πάρα πάρα πολύ μικρό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερη χρηματοδοτική υποστήριξη και πρέπει να αναγνωριστεί η αξία των ε, αγροτικών κοινοτήτων, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς. Χθε συζητούσαμε τα θέματα που προβληματίζουν την ε, παραγωγή γάλακτος. Αναγκάζονται οι αγρότες να ψάχνουν να βρουν και άλλες πηγές εισοδήματος. Τι θα γίνει όμως με τα εδάφια αυτά. Ποιος θα φροντίσει τα εδάφια αυτά, τις γέες αυτές. Ή θα τα αφήσουμε να επιστρέψουν στην κατάσταση που ήταν προ ετιών. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη δυνατότητας αποκόμισης κέρδους. Το βλέπουμε. Βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γαλακτοπαραγωγοί μας. Είπα εγώ και πριν ότι έχω μιλήσει με αγρότες ε, ε, λαμβάνονται αποφάσεις εδώ στις ε, Βρυξέλλες για το ηλεκτρονικό μαρκάρισμα των προβάτων και αυτό θα αναγκάσει πολλούς γεωργούς, πολλούς ε, αγρότες, συγγνώμη, να σταματήσουν την ε, κτηνοτροφία, την προβατοτροφία και να ασχοληθούν με άλλα πράγματα. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά. Είπατε και κάτι άλλο για το Access 3. Είναι εξαιρετικά αυτά. Αλλά πρέπει να δοθεί δυνατότητα στις εκμεταλλεύσεις και στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Ορισμένα από τα μέτρα που λαμβάνετε εμποδίζουν τους αγρότες από το να διαφοροποιηθούν, να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους. Ξέρω ότι θέλουμε την επικουρικότητα και όλα αυτά και εγώ είμαι υπέρ, αλλά υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου οι εθνικές κυβερνήσεις ή και οι ε, περιφερειακές διοικήσεις ξεφεύγουν από την πορεία και εκεί χρειάζεται να τους υπενθυμιστούν, υπενθυμιστούν τα πράγματα που είναι απαραίτητο να γίνουν. Μιλήσατε για 600 εκατομμύρια που πρόκειται να δαπανηθούν φέτος, που είναι δηλαδή προορισμένα για να δαπανηθούν. Οι κυβερνήσεις είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να καταθέσουν προτάσεις, βρισκόμαστε ήδη τον Σεπτέμβριο, μας μένουν ούτε τρεις μήνες ακόμη. Είμαστε σε θέση να απορροφήσουμε τα χρήματα αυτά ή θα χαθούν και πάλι τα κονδύλια αυτά και δεν θα φτάσουν ποτέ στους ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές περιφέρειες και που τα έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ, Τζέιμς. Μετά τη συζήτηση βεβαίως θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Χριστίνα Μόρδο. ezeket a hatalmas összegeket eh,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 I'm Ευχαρίστως να μιλήσω αγγλικά εάν διευκολύνω κάποιους. Καλά, καλά, θα τα πω στα αγγλικά. Φαίνεται πως ε, δεν ε, υπάρχει ε, μετάφραση από τα ουγγρικά, φαίνεται για κάποιο λόγο. Ζητώ συγγνώμη από τους Ούγγρους ψηφοφόρους μου που με παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, αλλά θα μιλήσω αγγλικά. Έχοντας δει αυτή την θαυμάσια παρουσίαση με τους ευγενείς στόχους, Διακόπτει ο πρόεδρος. Μπορείτε να μιλήσετε αν θέλετε στη μητρική σας γλώσσα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα σας παρακαλώ Κριστίνα. Ε, Για τους στόχους που ακούσαμε είναι σίγουρα πάρα πολύ καλοί. Οι αρχές είναι επίσης πάρα πολύ καλές. Πιστεύουμε ότι η Ήπεθρος ανθίζει Ακούμε ότι οι αγρότες ζουν μέσα σε ένα παράδεισο, αν πιστέψουμε όλα αυτά που ακούσαμε. Δεν είναι αλήθεια όμως, τουλάχιστον στη δικιά μου τη χώρα, σίγουρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το αντίθετο ισχύει. Οπότε, πού πάνε όλα αυτά τα ποσά, όλα αυτά τα χρήματα, τα κονδύλια, πού πάνε. Αυτό θέλω να ρωτήσω την ομιλήτρια. Ποιος είναι ο μηχανισμός ελέγχου που υπάρχει, που πανε αυτο θελω να ρωτησω την ομιλητρια ποιο ειναι ο μηχανισμος ελεγχου που ισχύει τι μέσα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ζητάει από τα κράτη-μέλη λόγο για τη χρήση των κονδυλίων. Αν πάντως τα χρήματα αυτά πηγαίνανε τελικά σε ευνοιοκρατία, σε δίκτυα μη ελεγχόμενα, αλλά όχι στις τσέπες των αγροτών, πώς θα μπορούσαμε να το ξέρουμε αυτό. Και τι θα έκανε σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σε θέση να παρακολουθήσει πού πάνε αυτά τα κονδύλια. Είναι σε θέση να επαληθεύσει ότι τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται πραγματικά για τους στόχους που καθορίστηκαν για αυτά. Θέλω λοιπόν μία απάντηση. Πώς ελέγχεται τα ποσά αυτά, πώς επαληθεύεται ότι δεν γίνονται καταχρήσεις και ότι δεν εξαφανίζονται τα χρήματα αυτά. Και μια άλλη ερώτηση. Πώς μπορούμε να κάνουμε την κοινωνία των πολιτών ε, να συμμετέχει, τις οικογένειες, τους ε, αγρότες, τις διάφορες επαγγελματικές οργανώσεις, τις οργανώσεις επίσης γυναικών τη υπαίθρου αγρότησών. Πώς όλοι αυτοί μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις για τη δαπάνη των κοδηλίων αυτών. Μέσα σε μια δημοκρατία, εγώ νομίζω ότι είναι οι εκλεγμένοι βουλευτές που έχουν αυτό το σκοπό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς διασφαλίζει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών όταν πρόκειται μάλιστα για τόσο μεγάλα ποσά. Ευχαριστώ. Μάρτιν Χόσλινγκ. Äh, Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι τα προγράμματα αυτά είναι σημαντικά για την μελλοντική εξέλιξη της γεωργίας. Είναι κρίσιμα και γι' αυτό μας ενδιαφέρει να λάβουμε και εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των προγραμμάτων. Είναι ωραίες και ευγενείς οι ε, φιλοδοξίες αυτές και οι στόχοι. Διερωτώμε όμως εάν όντως τα χρήματα αυτά πρόκειται να δαπανηθούν με σωστό τρόπο. Αυτό που βλέπω να λείπει, για παράδειγμα, είναι ένα κριτήριο δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. Έχουμε λοιπόν αυτά τα ωραία προγράμματα για δίθεν την αύξηση τη ανταγωνιστικότητα των αγροτών, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, έχει όμως νόημα να προωθούμε, να αναπτύσσουμε τις μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και να ε, αποδυναμώνουμε και να οδηγούμε σε ε, κατάργηση τις μικρές. Πού βρίσκεται εκεί η προσπάθεια δημιουργίας απασχόλησης, ιδιαίτερα για την γαλακτοπαραγωγή. Μπορούμε στην πραγματικότητα να προωθούμε μια πολιτική που αυξάνει την παραγωγικότητα, άρα και τις παραγόμενες ποσότητες, ενώ ήδη έχουμε πρόβλημα με την πλεονασματική παραγωγή. Είναι λοιπόν σωστή η στόχη αυτή. Μήπως εξακολουθούμε να προάγουμε την αύξηση της παραγωγής εν τέλει. Και το άλλο θέμα. Γιατί προωθείται η χρηματοδότηση μέσω τέτοιων προγραμμάτων ενός ευρέως φάσματος ε, παραγωγής, υποδομής της παραγωγής. Αυτά είναι, είναι ε, καθήκον προγραμμάτων συγκυρίας. Με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να γίνει. Πρέπει λοιπόν να επανελεχθεί η σκοπιμότητά τους. Τρίτο ερώτημα. Έχω την εντύπωση ότι οι νέοι στόχοι που διατυπώθηκαν Πάλι εδώ πρέπει να υπάρχει και το κριτήριο τη αντιμετώπιση τη αλλαγή του κλίματο. Η εντύπωσή μου είναι ότι στι χώρε μέλη τα προγράμματα εφαρμόζονται εν τέλει πολύ μέτρια. Δηλαδή, ναι, μεν οι στόχοι είναι υψηλή και φιλόδοξοι, στην πραγματικότητα όμω δεν αποδίδουν. Για παράδειγμα, περιορισμός των καλλιεργειών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του κλίματος δαπανώνται εδώ σωστά τα χρήματα ή απλώς στην πραγματικότητα οδηγούμαστε σε ενίσχυση κλασικών προγραμμάτων με τους κλασικούς παραδοσιακούς στόχους. Σας ευχαριστώ Μάρτιν. Σμιτ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Άκουσα τον συνάδελφο και εγώ Καλωσορίζω τους συναδέρφους από την Βόρεια Ιρλανδία. Ε, ως Σκοτσέζοι είμαστε πολύ κοντά. Να συνεχίσετε τη συνεργασία μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω επίση και τους συναδέρφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθαν εδώ. Ήμουνα στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης την προηγούμενη θητεία, τώρα ήρθα εδώ και ξέρω ότι υπάρχει συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα δύο. Επίσης, Πρέπει να σας πω ότι με απασχολεί το, το θέμα του προπολογισμού για την ανάπτυξη της υπαίθρου και την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι πολιτικές αυτές είναι εκείνες που βοηθούν οικονομικά τις περιοχές αυτές. Δυστυχώς όμως εμείς δεν έχουμε δικαίωμα απόφασης πάνω σε αυτό και να βλέπουμε τι γίνεται με το γαλακτοκομικό τομέα, πώς ε, οι παραγωγοί εγωπροβάτων εγκαταλείπουν τις δραστηριότητές τους, γιατί τελικά οι πολιτικές αυτές δεν αποφασίζονται εκεί που θα έπρεπε να αποφασίζονται. Δεν λέω ότι είμαι εχθρικός, αλλά θέλω να πω ότι φοβάμαι πως μερικές φορές υπάρχουν επικαλύψεις. Προσπαθούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Επικαλύπτονται αρμοδιότητες των κρατών μελών, με κίνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Ενώ αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι ότι είναι τα τρόφιμα. Ο κύριος στόχος της αγροτικής παραγωγής. Υπάρχουν νέες διαπραγματεύσεις στη Σκοτία για την ε, παραγωγή αγροτικών ε, προϊόντων. Είναι αλήθεια ότι υπήρξαν καταχρήσεις στο παρελθόν, ίσως γιατί τα κριτήρια δεν είχαν καθοριστεί αντικειμενικά. Και ακούστηκαν ανησυχίες και στη Σκοτία και τις έχω πει κι εγώ. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα για το τι κάνει η Επιτροπή για τα σχετικά κονδύλια από τον προπολογισμό. 600 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε όλοι τα θέλουμε. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη τι κάνουν για να διασφαλίσουν ότι θα δαπανηθούν αυτά τα χρήματα και πώς. Σίγουρα, αν υπάρχουν περιθώρια, με πάση περιπτώσει πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το ο κύριος στόχος της ε, αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τρόφιμα, παραγωγή τροφίμων, τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Bene, Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου μια ερώτηση. Ποιες <clears throat> διαφορές υπάρχουν μεταξύ των στόχων ανάμεσα στις παλές και στις νέες χώρες μέλη. Δηλαδή, οι χώρες που εντάχθηκαν το 2004 και 2007 έχουν την ίδια αναλογία 50-50 μεταξύ ε, των δύο πυλώνων ενώ οι παλές χώρες από ό,τι ξέρω είναι στο 17% για το δεύτερο πυλώνα. Και δεύτερο, βρίσκω θαυμάσιο να μιλούμε για περιφερειακή διαφοροποίηση, ότι υπάρχουν 88 προγράμματα. Έχουμε πράγματι πολύ διαφορετικές γεωργίες στην Ευρώπη και οι διαφορές βάθυναν ακόμα περισσότερα μετά από την ένταξη. Έχουμε την γεωργία που κατευθύνεται, προσανατολίζεται ανατολίζεται περισσότερε αγορές και εκείνη που έχει πιο πολύ κοινωνικό χαρακτήρα και που ε, στοχεύει σε μια <clears throat> περιφερειακή ανάπτυξη. Πώς μπορούμε αυτά να τα βάλουμε σε ένα κοινό παρονομαστή, δηλαδή αφενός ανταγωνιστικότητα στις παγκόσμιες αγορές, ποια, ποιους μηχανισμούς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκεί. Και ταυτόχρονα μια ενίσχυση των μικρών εκμεταλλεύσεων που έχουν πιο κοινωνικό χαρακτήρα ή σε περιφέρειες όπου η γεωργία καλείται να λειτουργήσει υπό δύσκολες συνθήκες και υπό η παραγωγή είναι μικρή, πώς μπορεί να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά της εν ώψη των παγκόσμιων αγορών. Εν προκειμένου και το μπορούμε να προωθήσουμε και το κριτήριο της καινοτομίας. Μιλούμε συχνά για ε, καινοτομία. Με ποιο τρόπο μπορούμε να την ενισχύσουμε. Πότε θα αρχίσει η συζήτηση περί προτεραιοτήτων και πολιτικών στόχων μετά από το 2013. Είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Ποιο είναι το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν προκειμένου. Και ε, ποια θα είναι η μοίρα του δεύτερου πυλώνα. Θα ενταχθεί στην κοινή αγροτική πολιτική ή στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Είναι μια συζήτηση η οποία διεξήχθη μεταξύ των επιτρόπων Φίσλερ και Μπαρνιέ. Αυτά θα τα ξαναδούμε. Γνωρίζουμε ότι πολλοί εμπειρογνώμονες και στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής συνηγορούν υπέρ της ένταξης του δεύτερου πυλώνα στην περιφερειακή ανάπτυξη. Και γνωρίζουμε επίσης ότι στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης η Ήπεθρος τελικά μειονεκτή. Βρίσκεται δηλαδή πάντοτε σε μειονεκτική θέση. Ευχαριστώ. Αντιπρόεδρος Νικολέσκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βασική μου μέρημνα είναι να δούμε πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε τα διάφορα εθνικά σχέδια αγροτικής ανάπτυξης. Πώς μπορούμε να βρούμε ισορροπία με άλλα λόγια μεταξύ δαπανών του άξονα 3 των υποδομών και του άξονα 1, αντιγωνιστικότητα. Ένα παράδειγμα. Το δικό μας εθνικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια για τις υποδομές που καλύπτουν σχεδόν όλο το ποσό που διατίθεται μέχρι το 2013. Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, τα προγράμματα που υπευλήθησαν είναι πάρα πολλά. Εκατοντάδες. Χρειαζόμαστε υποστήριξη για να μπορέσουν να ε, επιζήσουν οι εκμεταλλεύσεις. Όμως οι δικαιούχοι δεν έχουν διαφερθεί επαρκώς. Τα κράτη-μέλη λοιπόν πώς μπορούν να δώσουν όλα αυτά τα ποσά σωστά. Πώς μπορεί να υπάρχει ένας δοντολογικός κώδικας για να υπάρξει η μέγιστη αποτελεσματικότητα έναν οδηγό ορθής πρακτικής. Πρέπει να βρούμε καινούριε προσεγγίσεις. Ε, πρέπει να αποφύγουμε εγκατάλειψη εκμεταλλεύσεων αν απομονωθούν κάποιες περιοχές υπαίθρου. Θα πρέπει να διωθούν οι σωστές πρακτικές, να ενημερωθούν οι αγρότες, να ακολουθηθεί σωστή προσέγγιση. Αλλιώ δεν θα φτάσουμε πουθενά. Ευχαριστώ, Νίκο. Όλεκ Νίτσκακ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω μία παρατήρηση. Στην φάση προετοιμασίας των προγραμμάτων πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στην πρόθεση αυτής της ανάπτυξης, έτσι ώστε η ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου να βελτιωθεί. Κυρίως για εκείνους οι οποίοι ζουν σε μικρές γεωρικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό με ενδιαφέρει είναι τι απολογισμό μπορούμε εν να επιτύχουμε σε μια προοπτική λίγων ετών όπου λειτουργούν τα προγράμματα αυτά. Τι θέλουμε να πετύχουμε δηλαδή στις διάφορες χώρες, θέλουμε, ποια στοιχεία θέλουμε να διατηρήσουμε με ποιον τρόπο θα αλλάξουν οι εκμεταλλεύσει αυτές. Και κάτι που με ενδιαφέρει ακόμη είναι τι γίνεται μέσα στα πλαίσια αυτών των εκμεταλλεύσεων. Δηλαδή η πολιτική αυτή δεν πρέπει να αφορά μόνο τον αγρότη που είναι σήμερα 40, 50, 60 ετών, αλλά ποια θα, πώς θα επηρεάσει η πολιτική αυτή και την επόμενη γενιά αγροτών θα τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν την γεωργία ή θα παραμείνουν εν τέλει στην Ήπεθρο αλλά θα παραμείνουν τότε χωρίς απασχόληση. Ποιες ή πόσες θέσεις απασχόλησης μπορούμε να δημιουργήσουμε. Ασφαλώς η γεωργία είναι κάτι παραπάνω από την παραγωγή Δεν μιλούμε μόνο για αυξή του εισοδήματο του αγρότη. Χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Κάτι που οφείλει να μας ανησυχεί και εγώ το κρίνω διαφορετικά το αποτέλεσμα αυτό από, άλλοι, από άλλους συναδέλφους είναι πώς θα δαπανηθούν τα κονδύλια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αλλάζει ολόκληρη η δυναμική. Δηλαδή, <clears throat> πρέπει να φροντίσουμε να απορροφώνται τα κονδύλια ώστε να τον συντομότερο. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνο να πέσουμε σε μια παγίδα, όπως είδαμε για την γαλακτοπαραγωγή. Για την φάση 2007-2013 έχουμε επιτύχει απορρόφηση, αλλά μειώνονται οι τιμές. Προτιμώ να ασκήσουν κάποια πειθαρχία οι χώρες μέλη, να δώσουν περισσότερα χρήματα στην ανάπτυξη της περιφέρειας, για την παιδεία, για την βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και να προκαλέσουν μια αλλαγή νοοτροπίας, την οποία χρειαζόμαστε στην Ήπεθρο, ώστε η νέα γενεά να μην επαναλάβει τα σφάλματα των προηγουμένων. Ευχαριστώ. Τζοβάνι Λαβία Γκάτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση αυτή, αν και αντικειμενικά τη βρίσκω παροχημένη. Η παρουσίαση στο πρώτο τμήμα διηγήθηκε την τοποθέτηση όσον αφορά το προγραμματισμό 2007-2013, τίποτα όσον αφορά την ουσία της υλοποίησης των μέτρων. Δεν έχουμε επίκαιρες πληροφορίε όσον αφορά το επίπεδο αναλήψεως υποχρεώσεων, πληρωμών για τον προγραμματισμό. Αν μιλάμε για στοιχεία που έχουν μείνει δύο χρόνια πίσω, θέλουμε τώρα να ξέρουμε αντικειμενικά, τώρα που έχουμε γενικευμένη κρίση του αγροτικού συστήματος, τώρα που οι πόροι προορίζονται για τον άξονα 1, θα χρησιμοποιηθούν δύσκολα διότι λείπει ιδιωτική συγχρηματοδότηση για την υλοποίηση των επενδύσεων μαζί με το δημόσιο τομέα. Θα ήθελα να ξέρω ποιο, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε όσον αφορά την χρήση των πόρων. Δεύτερον, ο παλιός προγραμματισμός 2000-2006, από ό,τι σημείωσα, στις 30 Ιουνίου 2009 οδήγησε στην επικύρωση των δαπανών. Πώς πήγε η παλιά, ο παλιός προγραμματισμός. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το best practice. Ποιο θετικό πράγμα διαπιστώθηκε ότι πετεύθη. Και σε σχέση με τον προγραμματισμό, το επίπεδο επίτευξης των στόχων, ποιο είναι. Θα ήταν χρήσιμο να τα γνωρίζουμε όλα αυτά και θα ήμουν ευγνώμων στην στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορούσε να μας δώσει επαρκείς πληροφορίες. Ευχαριστώ και Τζοβάνι Λαβία. Ο κύριος ε, Σάντος. Ευχαριστώ, ο κύριο Καπούλα Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω κάτι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συστηματικά και σύντομα μας έδωσε τις πληροφορίες που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, καλό θα ήταν στην αρχή της θητείας που ξεκινάει τώρα, να ξέρουμε ότι εμείς έχουμε τεράστια ευθύνη Οπότε οι πληροφορίε αυτέ είναι για μια, μας για μια μεγάλη ευκαιρία. Καλό θα ήταν να μην ξεκινάμε με υποψίες σε βάρος των αγροτών ή των δικήσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχει το Λεκτικό συνέδριο που ήρθε εδώ εξάλλου χτες. Και έτσι νομίζω ότι δεν πρέπει εδώ να εκφράζουμε ανησυχίες και υποψίες για το πού πάνε τα χρήματα. Αν υπάρχουν συγκεκριμένες υποψίες και υπόνοιες, ας κάνουμε καταγγελία συγκεκριμένη στους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο. Εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξέρουμε ποιο είναι το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής στην πράξη να ξέρουμε τι έγινε με την ΚΑΠ μέχρι τώρα, ώστε να προσαρμόσουμε τη νέα ανάλογα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ο κόσμος όταν μας ψήφισε να δούμε κατά πόσο αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατίθεται τα κονδύλια. Ελπίζω κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής να βρούμε αρκετούς σύμμαχους ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε σε ένα νέο τρόπο εκπόνησης πολιτικής στον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου, όπου οι δικαιούχοι να είναι οι αγρότες. Όπως είπε και ο κύριος και πριν από λίγο, το σημερινό μοντέλο είναι τέτοιο όπου οι διάφορες ζώνες έχουν σαν αποτέλεσμα επικάλυψη της γεωργίας με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το μπέρδεμα. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσω τις ιδέες μου κάποια στιγμή, αλλά αυτό που ακούσαμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ορίσουμε το μοντέλο που θέλουμε στο μέλλον. Βάσει και τις εμπειρίες μας από το παρελθόν. Um, Κύριο Κέλλη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την έξοχη παρουσίαση. Πάρα πολλές λεπτομέρειες εμπειρία και πρέπει να ενημερωθούν τα στοιχεία μας αρκετά σύντομα. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Θα ήθελα να καλωσορίσω τα μέλη του Κοινοβουλίου της Βόρειας Ιρλανδίας σαν Ιρλανδός Ευρωβουλευτής από το Μάνστα την μεγαλύτερη αγροτική περιοχή της χαιρετίζω. Έχω ερωτήσεις. Πρώτον, αφορά το δεύτερο πυλώνα. Συμφωνώ με τον κύριο Νίκολσον, με πολλά από αυτά που είπε. Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε αυτά που υποθήκαν. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ θεωρίας και συνεπειών και αντιχτύπου. Ο πυλώνα λειτουργεί θεωρητικά, λογικά, όσον αφορά τα αποτελέσματα, τα επιτόπια. Περιορισμένα τα αποτελέσματα, λόγω του, επίπεδου χρηματοδότηση Και για του ντόπιου, για του γεωργού του κατοίκου τη υπαίθρου, πώ να του πείσουμε ότι θα αποκομίσουν ωφέλη. Αυτό είναι πρόβλημα. Κάτι άλλο που αντιμετωπίζουμε. Και το πιο σημαντικό που αντιμετωπίζω εκεί που ζω και από εκεί που κατάγομαι Πρέπει να είμαστε πιο προοδευτικοί στην καταπολέμηση των συνεπειών τη αυξημένη βιομηχανοποίηση τη γεωργία και το ίδιο ισχύει για τι οικογενειακέ εκμεταλλεύσει. Έχει τεράστιε κοινωνικέ συνέπειε αυτό. Από, την, από το Μόνστερ, από τη Νότια Ιρλανδία, το νότιο τη Ιρλανδία, αυτό είναι το πρόβλημα. Η αύξηση τη βιομηχανοποίηση τη γεωργίας και ο κοινωνικό αντίκτυπο. Πώ μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τον κόσμο. Διότι γίνεται σοβαρό πρόβλημα ξεπερνά το θέμα της γεωργίας. Τεράστιο πρόβλημα είναι, πώς να σας το πω. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να δούμε πώς τα χρήματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν την καταπολέμηση απώλειας εργασιών στη Γεωργία. Πρέπει να εξεταστεί το θέμα των νέων γεωργών που θέλουμε να εξακολουθούν να εργάζονται. Είναι πρόβλημα γενεών στη Γεωργία, κυρίως ε, στην Ιρλανδία. Η διαδοχή της Γεωργίας δεν χρησιμοποιούμε παρκώ τα κατάλληλα εργαλεία να κρατήσουμε τον κόσμο στις εκμεταλλεύσεις και να επιτρέψουμε σε περισσότερους γεωκτήμονες να ε, χρησιμοποιήσουν τη γη τους. Τα ξέρω καλά αυτά. Πρέπει να δούμε τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να καταργηθούν οι φραγμοί, τα εμπόδια που επηρεάζουν τους γεωργούς όσον αφορά τον τρόπο που αλλάζουν τον τρόπο εκμετάλλευσης της, των, εκμεταλλε... Ε, της, ε, των αγροκτημάτων τους. Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τίθενται θέματα. Πρέπει να εξετάσουμε τις σωστές πολιτικές. Θέλουμε πολιτικές που επιτρέπουν επικοινομορφία στη Γεωργία. Ίσως και κυβερνήσεις κινούνται εντός των πλαισίων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και δεν ξεφεύγουν και πρέπει να εξεταστεί. Χρειάζεται μεγαλύτερη ποικιλομορφία για να μείνουν οι γεωργοί στις εκμεταλλεύσεις. Δεν έχει προτεραιότητα το ευρυζωνικό δίκτυο, αλλά έχει προτεραιότητα εν γέννη, αλλά έχει προτεραιότητα για την ύπεθρο. Δεν ακούει καλά διερμηνέας, λυπούμε, αλλά υπάρχουν παράστα από το τηλέφωνο του αγορητού. Λοιπόν, τέλος, χρειαζόμαστε ανάλυση των επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα 600 εκατομμύρια θα δαπανηθούν προοδευτικό τρόπο. Διαφορετικά, τι θα πω εγώ στον κόσμο στην Ιρλανδία και στην εκλογική μου περιφέρεια. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ. Η ανάπτυξη της υπαίθρου νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δυστυχώς όμως έχει πολύ κακή χρηματοδότηση. Θυμάμαι τη συμφωνία του Δεκεμβρίου του 2005, αλλά δυστυχώς τελικά ε, δεν στηρίχθηκε η συμφωνία αυτή επαρκώ για την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Όντω χρειάζεται σοβαρή πολιτική για την ανάπτυξη τη υπαίθρου, αλλά στι διάφορε οικονομικέ προσπάθειες που γίνονται πρέπει να γίνει προσπάθεια και από τα κράτη-μέλη, ώστε και αυτά να δώσουν χρήματα. Δεν φτάνουν οι άμεσε ενισχύσει, χρειάζεται σωστή χρηματοδότηση. Πιστεύω στην κοινή γεωργική πολιτική και πιστεύω ότι αυτή πρέπει να καλύπτει το στόχο μας που είναι να έχουμε τρόφιμα σε καλές τιμές και ασφαλή για τον κόσμο. Συνεπώς αυτή είναι ευθύνη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας αυτής που πρέπει να αναλάβουμε εν μάλιστα της συνθήκης της Λισαβόνας. Και το λέω αυτό για την σωστή χρηματοδότηση, γιατί μετά από την τελευταία αναθεώρηση που έγινε της ε, αγοράς για τα καπνά, είχαμε πει ότι κάποια χρήματα θα περνούσαν στην ανάπτυξη τη υπαίθρου από τη Γεωργία. Εγώ λοιπόν εδώ θέλω να ξέρω αυτά τα κονδύλια από τα καπνά από το 2010, πού ακριβώς θα πάνε. Πού θα πάνε τα χρήματα αυτά ακριβώς. Και δεύτερον, υπάρχει μεγάλη ανησυχία από πλευρά των περιφερειακών αρχών στην Ισπανία και από τα συνδικάτα των αγροτών, από τους αγρότες και κτηνοτρόφους, για τα προγράμματα Ανάπτυξη τη υπαίθρου στη χώρα μου, στην Ισπανία, γιατί υπάρχει καθυστέρηση τουλάχιστον τριών ετών. Ρωτώ λοιπόν, η καθυστέρηση αυτή η τριετής στην Ισπανία μπορεί να σημαίνει ότι τελικά θα χάσει τα κονδύλια η Ισπανία που προβλέπονταν για αυτό το σκοπό. Κυρία Γιούζο Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα μας είπε. Έχω όμως την αίσθηση ότι τελικά ένα ξαναζασταμένο πιάτο μας σερβίρουν. Πάλι τα ίδια ακούμε. Χωρίς να ακούμε λύσεις για τη χρηματοδότηση όπως είπε και η συνάδελφός μόλις τώρα. Και θέλω να προσθέσω και κάτι. Το θέμα της γεωργίας δεν είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου. Με την ανάπτυξη της υπαίθρου βέβαια έχουν ε, εκμεταλλεύσεις οι αγρότες ε, με τις οποίες μπορούν να δουλέψουν αξιοπρεπώς. Αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται. Γιατί τι γίνεται με τους αγρότες, απαιτούμε τόσα πράγματα από αυτούς όσον αφορά το περιβάλλον, ένα σωρό πράγματα που τελικά οι αγρότες δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί απέναντι στις άλλες χώρες της παγκοσμιοποίησης που γνωρίζουμε. Όλα αυτά που απαγορεύουμε εμείς εδώ στους δικούς μας τους αγρότες μας έρχονται απ' έξω. Γιατί ο δεν μας επιτρέπει να απαιτούμε από τους άλλους αυτό το οποίο απαιτούμε από τους εαυτούς μας. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα της γεωργίας και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγκρίναμε τον κανονισμό για τα παρασιτοκτόνα. Στη Νότια Ευρώπη πρέπει να αφήσουμε πολλές εκμεταλλεύσεις γιατί αλλιώ δεν θα έχουμε αρκετά προϊόντα για να τα χρησιμοποιήσουμε ως παρασιτοκτόνα. Οπότε ό,τι απαγορεύουμε εμείς εδώ σε άλλες χώρες, στο Μαρόκο ή αλλού γύρω από τη Μεσόγειο, τέτοια προϊόντα που εμεί εδώ απαγορεύουμε, τα φέρνουμε. Κάνουμε ζημιά και στη Γεωργία και σίγουρα δεν βοηθάμε και τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Γιατί τελικά μας έρχονται προϊόντα από τέτοιε χώρες τα οποία έχουν υποστεί ε, τέτοιους ψεκασμούς από προϊόντα που εμεί εδώ απαγορεύουμε. Ευχαριστώ, Ζωζέ Μποβέ. Ευχαριστώ. Άκουσα προσεκτικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι αλήθεια ότι ακούμε τέτοια πράγματα. Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα, αναδιάφρωση. Μα είναι πρόβλημα αυτό όταν οι ακροτικές εκμεταλλεύσεις εξαφανίζονται οι γαλακτοπαραγωγοί εξαφανίζονται με τεράστια ταχύτητα εξαιτία τη μείωση των τιμών. Και εσεί μα μιλάτε για ανταγωνιστικότητα. Ε, τι θέλετε, όταν θα μείνουν δύο αγρότε, εντάξει, θα υπάρχει ανταγωνιστικότητα μεταξύ του, γιατί ο ένα θα είναι πιο ανταγωνιστικό από τον άλλον. Μα αυτό περιμένουμε. Το θέμα λοιπόν τη ανταγωνιστικότητα σαν μοντέλο είναι ένα μοντέλο ξεπερασμένο σήμερα. Το θέμα σήμερα είναι μπορούμε να παράγουμε για να προσφέρουμε τρόφιμα στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Και το τελευταίο παράδειγμα που εγώ γνωρίζω είναι εκείνο της Αγγλίας, που έχει ένα γνωστό τύρι, το τσένταρ, το ξέρουμε εδώ και καιρό. Ε, λοιπόν, φέτος για πρώτη φορά είχαμε αύξηση εισαγωγών τσένταρ. Δηλαδή η Αγγλία δεν καταφέρνει να παράγει το δικό της το τυρί. Απίθανο, ε. Απίστευτο. Έτσι θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο ή θα κάνουμε μια επανάσταση τύπου Κοπέρνικου. Πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο λοιπόν, σημείο αναφοράς που μέχρι τώρα ήταν ανταγωνιστικότητα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πούμε ότι δεν θα υπάρξει ανάπτυξη της υπαίθρου άμα δεν υπάρχουν πια αγρότες. Αλλιώς θα πρέπει να αλλάξουμε την έρημο και να την κάνουμε παραγωγική. Αλλιώ θα γίνει τουριστικός χώρος όπως είναι σε διάφορα σημεία Ινδιάνη, σε κάποιες προστατευμένε προστατευμένες περιοχές που θα πηγαίνουν οι τουρίστες και θα τους κοιτάνε. Ταντέν. Πιστεύω ότι μετά από τόσο ακούσαμε, καταλαβαίνουμε ότι τελικά ζητάμε πολλά από το δεύτερο πυλώνα. Ζητάμε από το δεύτερο πυλώνα και να εφαρμόζει μέτρα αλληλεγγύης, ε, αυτό το κάνουμε για τις ορεινές περιοχές, για παράδειγμα. Ζητάμε επίσης από το δεύτερο πυλώνα να συμμετέχει στον εξοχρονισμό και στην ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων της γης και ζητάμε επίσης και να χρηματοδοτήσει και κοινωνικά μέτρα υπέρ της γεωργίας. Και για το περιβάλλον επίσης. Ακούσαμε για την ανάκαμψη ότι θα χρηματοδοτήσουμε και την ανάπτυξη του ψηφιακού. Ωραία. Πρέπει όμως από τον προπολογισμό της γεωργίας να πάρουμε τα χρήματα. Όταν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το νέο οικονομικό προγραμματισμό μετά το 2013, εκεί θα πρέπει να κάνουμε σοβαρές επιλογές. Ο προϋπολογισμός της γεωργίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου πρέπει να χρηματοδοτεί τέτοια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε αυτά τα χρήματα για ανάπτυξη αστικών περιοχών. Τελειώσαμε. Όχι, έχουμε άλλη μια παρέμβαση. Δες, Άλμπερτ Δες. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη για την ε, μικρή μου σύντομη απουσία. Είχα μια, άλλη ψηφοφορία, είχα μια ψηφοφορία μάλλον σε άλλη επιτροπή. Θα ήθελα να επανέλθω σε ορισμένα πράγματα τα οποία είπε ο συναδελφός μου εδώ μου κύριος Τάντα. 45% των δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού είναι απαραίτητα για την γεωργία. Αλλά αυτό που θα μας οδηγήσει η ανάπτυξη της υπαίθρου σε διάφορες χώρες μέλη είναι διαφορετικές. Αλλά και μέσα στις ίδιες τις χώρες μέλη είναι διαφορετική ε, η ανάπτυξη υπαίθρου ανά περιφέρεια. Στα, στη χώρα μου χρήματα για την περιφερειακή ανάπτυξη χρησιμοποιούνται και για την αναγέννηση των χωριών. Έχουμε χωριά με 70 ε, σπίτια που έχουν δύο γεωργικές εκμεταλλεύσεις και όταν γίνεται αυτή η αναμόρφωση των ε, χωριών τελικά βρίσκουν οι γεωργοί ότι δεν μπορούν να περάσουν με τα γεωργικά μηχανήματα μέσα από το χωριό πλέον. Δεν επιτρέπεται. Δεν μπορεί να είναι αυτός όμως ο χαρακτήρας και ο στόχος της ε, αναγέννησης των χωριών. Θα πρέπει να εξευρεθούν κονδύλια και από άλλες γραμμές του προϋπολογισμού ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ευρείας ζώνης υποδομή για ε, την Ήπεθρο, ώστε να λαμβάνονται και να υλοποιούνται μέτρα τα οποία πραγματικά να εξυπηρετούν την γεωργία. Νομίζω ότι υποστηρίζουν όλοι οι συναδελφοί μου εδώ ότι η καλύτερη ανάπτυξη της περιφέρειας θα βασιστεί σε μια σωστή ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής. Ωραία. Θα ήθελα, δίνοντας το λόγο στην κυρία Λόρις Χόφμαν, να αναφέρω κι εγώ κάποια πράγματα. Είναι ένα σημαντικότατος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής η ανάπτυξη της υπαίθρου. Κούσαμε σε όλε τι παρεμβάσει μια επιθυμία συγκεκριμένων στοιχείων, συγκεκριμένων πραγμάτων. Στο επίκεντρο να μπουν οι απαιτήσει των γεωργών μα. Συχνά βλέπετε στην Ευρώπη ασχολούμαστε με τι σωστέ ευαισθησίες των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά το περιβάλλον. Μιλήσαμε για τα παρασιτοκτόνα, για την καλομεταχείριση των ζώων τις νέες ευαισθησίες της σημερινής ε, κοινωνίας. Οι γεωργοί μας πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες. Όμως συχνά δεν δίνουμε την ίδια προσοχή σε αυτό που πρέπει να κάνουν μετά οι αγρότες για να συνεχίσουν να ζουν, να συνεχίσουν να επιβιώνουν, να είναι ανταγωνιστικοί, να παίζουν ρόλο στην αγορά. Πιστεύω λοιπόν ότι η προσπάθεια πρέπει να καταβάλουμε για την υποστήριξη του σημαντικού πυλώνα της αγροτικής πολιτικής, την ανάπτυξη της υπαίθρου, πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι στο επίκεντρο είναι η γεωργία. Αυτή είναι η σταθερή γεωργία που είπε ο Αλμπερντές. η γεωργία που θέλουμε να παίξει ρόλο ε, στην αγορά, όπως είπε ο Λουίς Καπούλα Σάντος. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε το στόχο της πολιτικής μας. Δηλαδή θέλουμε ισχυρή γεωργία που ζει και επιβιώνει στην παγκοσμιοποίηση. Ποτέ να λησμονούμε το ευρωπαϊκό αγροτικό μοντέλο για το οποίο είμαστε υπερήφανοι, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι οι γεωργοί μας θα πρέπει να ανταγωνιστούν άλλους, άλλες ισχυρές γεωργίες στον κόσμο. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο αμέσως στην ε, κυρία Χόφμαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις συζητήσαμε πολλές από αυτές. Τροφή προσκέψη για μας. Αναφερθήκατε σε πολλές πτυχές. Θα τις εξετάσουμε τους επόμενους μήνες, όταν θα εξετάζουμε το μέλλον. Καταρχάς, το οικονομικό κομμάτι. Ο κύριος Νίκολσον θεωρεί ότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο δεύτερο πυλώνα. Ισχύει σε κάποιο βαθμό αυτό. Θα ήταν παραπλανητικό να θεωρούμε ότι ακόμα και με το εντυπωσιακό βαθμό, τα 225 δις, μπορούμε να οργανώσουμε τα πάντα στην Ευρώπη και στη Γεωργία. Είναι για ένα μικρό κομμάτι των χρημάτων που απαιτούνται για τη γενική προσαρμογή, αναδιάρθρωση σε σχέση με τις υπάρχουσες οικονομικές απαιτήσεις για την Ήπεθρο. Να πω ότι αυτά που, που διαπιστώσαμε αυτή την περίοδο ήταν λιγότερα από τις προσδοκίες μας. Το αρχικό ποσό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπε η κυρία Γκαρσία, μειώθηκε με κάτι παραπάνω από 20 δις, περικοπή πάνω από 20 δις και κάτι άλλο. Ας ληφθεί υπόψη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα εμείς. Πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους και τα κράτη-μέλη. Μιλάμε για συνεργασία. Πρέπει τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα χρήματα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς από εδώ. Είναι ευθύνη των κρατών μελών να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα χρήματα. για τα 600 εκατομμύρια. Τα 600 εκατομμύρια από το πακέτο ανάκαμψης είναι ε, ανάληψη υποχρεώσεων πληρωμών, πρέπει να ενταχθούν στον προϋπολογισμό το φετινό, πρέπει να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν χρειάζεται να, να εκμεταφιεθούν φέτος. Δύσκολο να εγκριθεί ένα πρόγραμμα Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Ε, πότε θα πληρώσουν τα χρήματα, καταβάλουν τα χρήματα. Και στην ανάπτυξη πέθρου και σε όλα τα ε, ταμεία υπάρχει περιθώριο. Αναλαμβάνει μια δέσμευση, μπορεί να αποφασίσει για ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να προωθήσει. Τα κάτι μελη μπορούν ήδη να αδειοδοτήσουν, να αναλύσουν συγκεκριμένα προγράμματα. Αλλά μπορούν να καταβάλουν τα χρήματα τη διετία μετά την ανάληψη της υποχρέωσης. Μέχρι το τέλος του 2012 μπορούν να εκταμιευθούν και να καταβληθούν τα χρήματα. Δεν χρειάζεται να δαπανηθούν όλα σε ένα χρόνο. Κάτι τέτοιο θα ήταν ανέφικτο. Υπάρχει επαρκή έλεγχος της χρήση των χρημάτων. Ήταν ένα ερώτημα αυτό. Υπάρχει μια δομή που έχει αποφασιστεί όσον αφορά την πολιτική. Πάμε τώρα στις επίσημους ελέγχους. Τα κράτη με κανόνες που προβλέπουν οι κανονισμοί πώς πρέπει να γίνεται ο έλεγχος. Γίνεται διοικητικό έλεγχος, επιτόπιος έλεγχος επίσης. Να δουν κατά πόσο ε, ε, είναι σωστή επένδυση, αν πράγματι ο Γιώργος έχει τη δηλωθεί σε έκταση ή όχι. Αν ο Γιώργος κάνει αυτά που απαιτούνται ή και άλλοι που παίρνουν τα χρήματα, αν κάνουν αυτό που πρέπει. Αν οι δαπάνες συμφωνούν με τον κανονισμό. Όχι μόνο αν το ποσό είναι το σωστό ποσό, αλλά αν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά το ποσό. Γίνονται έλεγχοι γι' αυτό. Έχουμε ένα ελεγκτικό πλαίσιο λοιπόν. Αλλά και τα κράτη-μέλη πρέπει να υποβάλουν αναφορέ να μας πούν τι κάνουμε τα χρήματα. Στην ανάπτυξη υπαίθρου έχουμε αιτήσει εκθέσει. Τα κράτη-μέλη πρέπει να αναφέρουν την χρήση των χρημάτων, πώ χρησιμοποιήθηκαν, ποια τα αποτελέσματα τη χρήση των χρημάτων, δείκτες αποτελεσμάτων και δείκτες α, συνεπιών αντικτύπου πρέπει να υποβάλλονται. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Έχουμε κοινού δείκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε αυτή τη φάση. Έχουν συμφωνήσει και τα κράτη-μέλη. Όλα τα κράτη-μέλη αναφέρουν τα ίδια πράγματα. Και επίση και το επίπεδο απασχόληση, τη απασχόληση που δημιουργούνται. Αν έχουμε στοιχεία για την απασχόληση, έχουμε αριθμό δικαιούχων, ποσά που χρησιμοποιήθηκαν και ποιο περίπλοκους δείκτες για τον αντίκτυπο συγκεκριμένων πολιτικών όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων Φερρυπίν. Είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο από μόνο το αυτό. Τα κράτη-μέλη πρέπει να αναφέρουν κάθε χρόνο τι κάνουν και πρέπει να αναφέρουν δύο φορές κατά τη διάρκεια της περίοδου εάν έχουν πετύχει τους στόχους της στρατηγικής τους. Έχουμε στρατηγική έκθεση το 2010, υπάρχει και ενδιάμεση έκθεση που αφορά την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων των κρατών μελών. Πρέπει να πω όμως ότι δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολο να πάρουμε τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία από τα κράτη-μέλη, είναι περίπλοκο. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη σε επιτροπές. Έχουμε συγκεκριμένο δίκτυο αξιολογήσεως. Υποστηρίζουμε την προσπάθεια των κρατών μελών να μας ενημερώσουν για τα αποτελέσματα των πολιτικών, για τον αντίκτυπο των πολιτικών. Είναι σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό. Το τονίζουμε όλος ιδιαίτερος. Εν πάση περιπτώσει έχουμε στόχους που καθορίζονται από τα κράτη-μέλη. Εντάσσονται στα προγράμματά τους. Πρέπει να αναφέρονται στοιχεία για τους στόχους. Ποιε πρέπει να είναι συνέπειε των προγραμμάτων του, Ποια πρέπει να είναι τα αποτελέσματα διαφόρων μέτρων στι διάφορε περιοχέ και ποια είναι η εκροή δεν έχουμε τα στοιχεία από όλα τα κράτη-μέλη, αλλά έχουμε πλήρη στοιχεία για πάνω από 50 από τα 88 προγράμματα. Σας διαβεβαιώ όμως ότι είναι πολύ σκληρή δουλειά αυτή και τα κράτη-μέλη προσπαθούν να βελτιώσουν τα συστήματά τους. Πρέπει να ελέγχεται μία πολιτική για να είναι αξιόπιστη προς το κοινό. Εγώ παρουσίασα μια στατική εικόνα. Δεν σας είπα ακριβώς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνει αυτό τη στιγμή που θα γίνει ο αναπρογραμματισμός του ελέγχου υγείας και θα έχουμε καλύτερη εικόνα όσον αφορά το στάδιο εκτελέσεως της πολιτικής και θα επανέλθουμε σε αυτά. Ο κύριος Χολστάιν έθεσε το ερώτημα για τη, θέση, για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια της πολιτικής αναπτύξεως υπαίθρου. Σε κάποιο βαθμό δόθηκε από κάποιους συναδέλφου η απάντηση. Είπαν ότι όσον αφορά τη γεωργία παλεύουμε κατά της απώλειας θέσεων εργασιών. Δεν νομίζω να πιστεύει κανεί ότι θα δημιουργηθούν πολλέ θέσει εργασία, νέε θέσει εργασία. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, αλλά μέσω διαφορετική πολιτική από αυτή που επιδιώκουμε τώρα. Έτσι που έχουν τα πράγματα, μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε τον τομέα και αυτή η αναδιάρθρωση μπορεί να συμβάλλει στην διατήρηση θέσεων εργασία. Είναι θέσει εργασία που μπορούν να είναι βιώσιμε. Θέσει που μπορούν να αντισταθούν στις εξελίξεις στην αγορά, να κρατήσουν. Δύσκολο όμως κανείς όταν κινείται σε ανοιχτές αγορές και εκμεταλλεύσεις που ανταγωνίζονται μία την άλλη. Είναι δύσκολο. Τα μέτρα του άξονα 3, 3 αυτό προσπαθούν να κάνουν, δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ποια είναι η κεντρική ιδέα να στην ανάπτυξη υπαίθρου να υπάρχει μια συνιστόσα που αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Επενδύσεις για ευρυζωνικέ υπηρεσίε είναι κάτι που πρέπει να γίνει σχετικά γρήγορο. Δεν μπορούμε να το αναβάλουμε. Θα μου πείτε τι σχέση, έχει, τι σχέση έχουν οι ευρυζωνικέ υπηρεσίες με τη γεωργία. Οι περισσότεροι γεωργοί σήμερα έχουν έναν υπολογιστή προσωπικό, βλέπετε. Σχεδόν όλα τα λογιστικά τους βασίζονται στο διαδίκτυο. Και το ίδιο ισχύει και για εκείνους που ψάχνουν να πάνε για διακοπές σε ένα αγρόκτημα. Πρέπει και η οικογένεια του Γεωργού χρησιμοποιεί τον υπολογιστή. Έχουμε και κοινωνική διάσταση όσον αφορά τις ευρυζωνικές υπηρεσίες που θεωρούμε ότι είναι σημαντικές. Τώρα από πού θα έρθουν τα χρήματα, από αυτό το ταμείο ή από άλλο ταμείο, αυτό είναι άλλο ερώτημα. Πάντα όμω συμπεριλαμβάναμε αυτά τα μέτρα στην ανάψη πέθρου. Κατά το παρελθόν δίναμε προτεραιότητα στις παροχές υπηρεσιών και στην κατάρτιση. Συνεχή κατάρτιση για να μπορούν να μαθαίνουν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν την τεχνολογία, να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες. Οι υποδομές είναι θέμα διαθροτικών ταμείων Περιφερειακό, μιλάμε για περιφερειακό επίπεδο. 12 δις έχουν τα κατά ταμεία όσον αφορά τη δημιουργία υποδομών. Μόνο δύο από τα 12 δις δίνονται για δημιουργία υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών. Το πρόβλημα στην Ήπεθρο δεν υπάρχουν υποδομές. Πώς να παράσχεις υπηρεσίες ή κατάρτιση όταν δεν υφίσταται υποδομή, πώς θα χρησιμοποιήσεις μια μη υφιστάμενη υποδομή, θα μπορούσαν να εργαστούν τα ταμεία και να γίνει καταμερισμός εργασιών μεταξύ των ταμείων. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα πιέσουμε, να τα υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη, να δημιουργήσουν συγκεκριμένο μοντέλο χρηματοδότησης για αυτό το στόχο. Αυτό είναι η δική τους υπόθεση. Στα προγράμματα των κρατών μελών θα πρέπει να προβλέπεται η χρήση των ε, πόρων για συγκεκριμένους σκοπούς. Όσον αφορά κάτι άλλο που υπόθηκε, ο κ. Σμίθ νομίζω, είπε ότι ο μόνος στόχος που θα έπρεπε να κάνουμε είναι η παραγωγή τροφίμων που θα είναι επικερδής, να είναι ο μόνος στόχος για τη γεωργία. Είναι ένας από τους στόχους πιστεύω. Έχω την εντύπωση ότι η κοινωνία θέλει και άλλα πράγματα. δεν πρέπει να είμαστε κοντόφθαλμοι όσον αφορά το τι μπορεί να παράσχει η γεωργία. Θα είναι ένα είδος αυτοπεριορισμού. Αν πούμε πρέπει να παράγουν μόνο τρόφιμα, υγιή τρόφιμα σε χαμηλές αποδεκτές τιμές. Αν το πούμε αυτό θα αφαιρέσουμε πάρα πολλά από τη γεωργία. Πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Ε, χρησιμοποιεί πάνω από 90% των εδαφών η γεωργία ε, οι πολίτες θέλουν να συντηρηθεί το τοπίο, βασικά χαρακτηριστικά του τοπίου κλπ. Και κάποια περιβαλλοντικά ωφέλη που μπορεί να μα δώσει η γεωργία θέλουν οι πολίτες. Αν υπάρχει μια αγροτική παραγωγή πρέπει να είναι βάση για να παράγει δημόσια αγαθά όπως αποκαλούνται και άλλα συναφή δημόσια αγαθά. ετέσαν διάφορα θέματα που είναι περίπλοκα. Προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε τα όρια που έχουμε θέσει για τις, λιγότερο, για τις περιοχές που είναι σε δυσμενή θέση και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Έχουμε ενδιάμεση κατηγορία εκεί που υπάρχουν φυσικά προβλήματα, ελαττώματα που αυξάνουν το κόστος για τους γεωργούς γιατί είναι σε δύσκολες περιοχές και πρέπει να τους βοηθήσουμε να ανταγωνιστούν για να μην εγκαταλείψουν την γη τους. Αυτό είναι κάτι που τα αναφέρατε επανειλημμένα. Υπάρχει ένας κίνδυνος πράγματι στις περιοχές που είναι περιθωριακές, δύσκολες. Οι γεωργοί να μην θέλουν να μείνουν, αλλά τους συμφέρει. Δεν θέλουν να καλλιεργούν τις εκτάσεις εκεί και αυτό αν γίνει θα είναι πρόβλημα για τη βιοπικιλότητα, αλλά και για, την, για τον κοινωνικό ιστό της περιοχής. Τώρα η διαδικασία των ορίων που θέτουμε είναι κάτι δύσκολο. Θέλουμε να είναι σύστημα διαφανέστερο, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Εφαρμόσιμο σύστημα και στα 27 κράτη-μέλη, βάσει δικτών. Το εξετάζουμε, το συζητούμε με τα κράτη-μέλη το θέμα και τα κράτη-μέλη προσπαθούν επιτεχνικής τεχνικής να δουν κατά πόσο ένα συγκεκριμένο σύστημα του κοινού, του μεικτού κέντρου ερευνών του ΙΣΠΡΑ, το μοντέλο αυτό που έχει χρησιμοποιηθεί. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να μας πούν τι θεωρούν, τι πιστεύουν. Τι έγινε με τις προσωμιώσεις και με τις δοκιμές που έκαναν. Κεντρική ιδέα είναι ότι έχουμε 150 διαφορετικούς δείκτες τώρα που χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη για να καθορίσουν αυτές τις περιοχές. Αν καταφέρουμε να μειώσουμε τους δείκτες και να τους εναρμονίσουμε, τότε βελτιώνεται η αξιοπιστία του συστήματος και μπορούμε καλύτερα να βλέπουμε πώς λειτουργεί και να προσμετρούμε τα αποτελέσματα. Το θέμα της ανταγωνιστικότητας, ένα άλλο θέμα που εφήγει ο κ. Μπουφέ το έθιξε. λέμε πάντα ότι οι άνθρωποι να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, πρέπει να προοδεύσουν κλπ. Τα χρησιμοποιούμε σαν συνθήματα. Ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να περιγραφεί πολύ σύντομα. Μπορεί να έχει μια πολύ μικρή εκμετάλλευση και να είσαι ανταγωνιστικό. Αλλά δεν μπορεί να είσαι μικρή εκμετάλλευση, να έχει δύο εκτάρια στάρι και πέντε βόδια και να επιβιώσει. Το θέμα της ανταγωνιστικότητας πώς τίθεται, πώς μπορούν να επιβιώσουν οι γεωργοί, πώς μπορούν να ζουν στις παρούσες περιστάσεις, να κάνουν τη δουλειά τους. Και τα κράτη-μέλη θα προσπαθήσουν να προτείνουν κάποιες δυνατότητες στους γεωργούς. Πώς να προσαρμοστούν, να σκεφτούν διάφορους τρόπους για βιολογικές καλλιέργειες Φερρυπίν, ας μην πούμε σε λεπτομέρειες τώρα, οι βιολογικές καλλιέργειες, οι γεωργοί που ασχολούνται με βιολογικές καλλιέργειες είναι ανταγωνιστικοί. Δεν είναι ότι έχουμε μεγάλες εκμεταλλεύσεις και μικρές που δεν είναι εκμεταλλεύσεις ανταγωνιστικές. Δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ του τι είναι μικρό, τι είναι μεγάλο. Αν σε μία πολιτική δεν θεωρήσουμε ότι δεν πρέπει να κινηθούν προς μία κατεύθυνση οι γεωργοί για να επιβιώσουν, Δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, αλλά να το συνειδητοποιήσουν οι ίδιοι. Δύσκολο τώρα μια πολιτική να προστατεύσει τον κόσμο, τους γεωργούς, από τα πάντα. Από προβλήματα που έρχονται από τις αγορές και από εξωτερικούς παράγοντες. Ανταγωνιστικός δεν σημαίνει πάντα μεγάλες μονάδες, αυτό θέλω να πω. Δεν σημαίνει ότι θα, θα εξαφανιστούν οι μικρές εκμεταλλεύσεις. Κάτι που αναφέρθηκε πρέπει να πούμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε περίπου 6 περίπου εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη. Εκμεταλλεύσεις που δεν μπορούν να ζουν από τη γεωργία, άλλου είδους εκμεταλλεύσεις. Έχουν δύο δυνατότητες. Ή κάνουν το άλμα αυτά τα 6 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις και γίνονται πιο παραγωγικές εκμεταλλεύσεις και επιβιώνουν μέσω της γεωργίας ή αυτές οι εκμεταλλεύσεις ε, βρίσκουν άλλες δυνατότητες για να επιβιώσουν οικονομικά. Και θέλουμε να τους δώσουμε δυνατότητες που μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη και κυρίως μέσω της ε, των δραστηριοτήτων. Δηλαδή γεωργοί που δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνο από τη γεωργία ή θέλουν να κάνουν κάτι άλλο, να δημιουργήσουν άλλες επιχειρήσεις, αυτοί οι γεωργοί να τύχουν υποστήριξης. Μέχρι τώρα το 13% των χρημάτων από αυτό το κονδύλι που δεν πηγαίνει κατευθείαν στη γεωργία. Είναι το ποσοστό που δεν πηγαίνει κατευθείαν στη γεωργία, πάντα το ξέρουμε αυτό. Λέμε η πολιτική ανάπτυξη υπαίθρου παίρνει τα χρήματα της γεωργίας. 30% πάει στον άξονα 3. Μεγάλο ποσοστό πάει για την ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων των γεωργών. Να βάλουν πόδι και σε άλλη δραστηριότητα. Αυτό προσπαθούμε να του βοηθήσουμε. Μεταφορές, Φερρυπίν. Ασχοληθούμε με μεταφορές. Να μπουν στο τουριστικό τομέα. Και ούτω καθεξής. Και αυτό που είναι, είναι εκτός γεωργίας αυτή η δαπάνη. Μικρό ποσό είναι αυτό. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις τα χρήματα πάνε στη γεωργία. Άμεσα στη γεωργία. Εάν πάνε άσχημα τα πράγματα, αυτά και γίνουν αυτά που είπε και ο κ. ότι επειδή έχει ανακαινιστεί ένα χωριό δεν μπορούν να περάσουν με τους γεωργικούς ελκυστήρες οι γεωργοί πλέον από τα τρακτέρ τους. Αυτό είναι άλλο θέμα. Με ρωτήσατε πώς πώς, μπορεί, πώς μπορούν αυτοί που εργάζονται στην διοίκηση να επηρεάσουν την πορεία των χρημάτων. Έχουμε την Επιτροπή Παρακολούθησης. Να. Επιτροπή Παρακολούθησης για κάθε πρόγραμμα. Όλοι εκπροσωπούνται και όλοι οι εμπλεκόμενοι. Περιβαλλοντικές ομάδες. Περιφερειακές ομάδες. Εκείνοι που θα προστατεύσουν το περιβάλλον και τα τοπία συμπεριλαμβάνονται. Τα υπουργεία συμπεριλαμβάνονται. Οι πάντες. Όλοι αυτοί έχουν λόγο σχετικά με το τι γίνεται με το πρόγραμμα. Και κάτι άλλο. Έχουμε τον κανονισμό. Λέμε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έρθονται σε διαβούλευση με τους εμπλεκομένους όταν ετοιμάζουν το πρόγραμμα ή όταν επιφέρουν μια σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα. Είναι προϋπόθεση αυτή, όρος. Πρέπει να δούνε ποιες είναι οι απόψεις των εμπλεκομένων, ποια είναι τα συναισθήματά τους, ποιες είναι οι ανάγκες τους, τι πιστεύουν. Αλλά αυτή είναι η γενική προσέγγιση, γενικός τρόπος διοργανώσεως μιας διαδικασίας. Μέσω του leader μπορεί να υπάρξει ο μεγαλύτερος επηρεασμό και γι' αυτό προωθήσαμε και προωθούμε αυτή την προσέγγιση. Διότι θεωρούμε ότι οι ντόπιοι πρέπει να έχουν λόγο για αυτά που γίνονται σε μια περιοχή. Συμφωνώ βέβαια ότι η κατάρτιση και η διάδοση βελτίστων πρακτικών είναι σημαντικότατο ζήτημα. Το λέμε στα κράτη-μέλη αυτό. Διότι υποτιμάται συχνάκης. Μπορεί να έχεις άριστα μέτρα, κυρίως αγροπεριβαλλοντικά, αλλά οι γεωργοί καμιά φορά δεν ξέρουν τι να κάνουν, ακριβώς τι να κάνουν. Και αυτό φορά και τη διαχείριση του νερού, των υδάτων, κρίσιμο θέμα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με το νερό στην Ευρώπη. Και οι γεωργοί πρέπει να έχουν δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβουλή, κάποια κατάρτιση, κάποια υποστήριξη. Πώς να τα καταφέρουν καλύτερα. Και τα κράτη-μέλη έχουν κάθε συμφέρον να καταβάλουν σχετικά μια προσπάθεια. Σχετικά με το ζήτημα. Και άλλο ερώτημα ετέθη. Ποια είναι η μορφή των δαπανών στα παλιά και νέα κράτη-μέλη, αν υπάρχει διαφοροποίηση. Υπάρχουν μικροδιαφορές. Η γενική εικόνα ίδια. Δηλαδή, στο δεύτερο άξονα πάνε τα περισσότερα χρήματα. Και στον άξονα 3 πάνε τα λιγότερα. Εν γέννη τα νέα κράτη-μέλη είναι ισχυρότερα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Άξονα 1. Βλέπουν ότι πρέπει να αναδιαρθρωθούν τώρα οι εκμεταλλεύσεις τους. Να ανταποκριθούν στις απαιτήσει της αγοράς. Δεν ασχολούνται τόσο με περιβάλλον. Ούτε με τον άξονα 3. Και καμιά φορά είναι λυπηρό αυτό διότι χρειάζονται οικονομικές δραστηριότητε στην Ήπεθρο και εκτός Γεωργίας προς όφελος μάλιστα των νέων που θέλουν να παραμείνουν στις περιοχές αυτές και δεν θέλουν να φύγουν αλλά τελικά μπορούν να μείνουν μόνο αν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν χρήματα και να δουλέψουν εκεί. Τέλος, η κυρία Γκαρσία είχε ένα ερώτημα όσον αφορά τι για τον καπνό και πώς σχετίζεται με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Τα κράτη-μέλη έχουν βάλει αυτά τα ποσά, έχουν πάρει στα αναψιακά τους προγράμματα κάποια ποσά. Κάποια κράτη-μέλη στην αρχή της περίοδου προγραμματισμού έχουν σαφή στατηγική, δηλαδή τι πρέπει να συμβεί στις διάφορες περιοχές. Αυτές που πλήττονται από τις αλλαγές στην αγορά όσον αφορά τον καπνό. Και είπαν ότι για κάποιες, καπνοπαραγω... κάποιες ποιότητες καπνού θέλουν να βελτιώσουν την κατάσταση. Και κάποιες καλλιέργειες δεν θα ήταν βιώσιμες στο μέλλον και θέλουν να προσφέρουν άλλες δυνατότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν πολλά μέτρα αναπτύξεως της υπαίθρου για να ενισχύσει κανείς ε, ή να κρατήσει μια παραγωγή που είναι βιώσιμη παραγωγή. Ούτω ώστε να επιβιώσει. Υπάρχουν πολλά εργαλεία και μέσα για εκείνου που θέλουν να εγκαταλείψουν τον τομέα και να κάνουν κάτι άλλο. Να ασχοληθούν με άλλη αγροτική παραγωγή ή αν αυτό είναι ανέφικτο σε κάποιε περιοχέ να βρουν αλλού απασχόληση εκτός γεωργία. Και υπάρχει δυνατότητα επίση οι μεταπητικέ επιχειρήσει να προσαρμοστούν αλλά υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη που δεν έχουν σαφή στρατηγική και τονίζουν έντονα την παροχή επενδύσεων στον τομέα του καπνού. Και αν δεν είναι σαφής ο στόχος των επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή της αγοράς, δύσκολο να κρίνει κανείς τα μέτρα και τα προγράμματα. Όπω ειπα είπα, υπάρχουν κράτη-μέλη που είναι προχωρημένα εκεί, ήδη κινούνται και άλλα κράτη-μέλη που είναι, πώ να το πω, δεν έχουν καταλήξει κάπου. Και περιμένουμε. Είμαστε σε επαφή με τα κράτη-μέλη αυτά. Εξετάζουμε τις προτάσεις τους. Και περιμένουμε να δούμε τι εξηγήσει θα μας δώσουν. Νομίζω ότι λίγο πολύ Απάντησα. Αν δεν απάντησα σε όλα, ζητώ συγγνώμη. Ελπίζω να έχουμε δυνατότητες και για άλλη ανταλλαγή απόψεων. Και με τα χαράς, μετά τον αναπρογραμματισμό, να έρθω να σας παρουσιάσω συγκεκριμένα στοιχεία. Οικονομικά στοιχεία μπορώ να σας δώσω για φέτος μόνο. Αυτό δεν είναι ικανοποιητικό βέβαια. Δεν είναι καλό να σας δώσω στοιχεία και για τους δικαιούχους, πού πηγαίνουν τα χρήματα, υπό ποιες συνθήκες κλπ. κλπ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστούμε την κυρία Λόρις Χόφμαν, Χόφμαν, ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα συνεχίσουμε σίγουρα και περιμένουμε κι άλλες ειδήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας πάμε εντάχει στα τελευταία δύο σημεία που έχουμε για να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας. Στο σημείο 13 αφορά την επιβεβαίωση του χρονοδιαγράμματος της Επιτροπής Γεωργίας για το 2010. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε λοιπόν το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα για το 2010. Το πρόβλημα είναι ότι ζητήσαμε ε, μέγιστε, συμμορφωτήκαμε τις μέγιστες απαιτήσει και ίσως τελικά να, να χρειαστούμε λιγότερο χρόνο από ό,τι προβλέψαμε. Σας ενημερώνω λοιπόν για το πρόγραμμα των, του επομένου χρόνου των εργασιών. Το πρωί συζητήσαμε τους συντονιστές των ομάδων. Πήραμε κάποιες αποφάσεις όσον αφορά τους εισηγητές και τις εκθέσεις και ως ήθιστε επικεφαλής των ομάδων θα σας ενημερώσουν δεόντως για τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Τέλος, στα διάφορα, ζητήσατε το λόγο, Στιουαρτ. Θέλετε το λόγο. Και με αυτή την παρέμβαση θα κλείσουμε τις εργασίες ε, των, της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε. Θέλω να πιστήσω την προσοχή της Επιτροπής όσον αφορά την κτηνοτροφία. Ο... Εμείς στο Norfolk με την εταιρεία χείριου κρέατος έχουμε διαπιστώσει ότι πουλάει με μια ζωτροφές με αύξηση πρωτεΐνης μέσα για να αυξήσει την παραγωγή. Πρώτη φορά στα 30 χρόνια λοιπόν ε, έχει ειδοποιηθεί ο κύριος Λόρενς ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η προμήθεια ζωτροφών σε αυτόν. Οπότε απειλείται η επιχείρησή του και οι λόγοι είναι καθαρά πολιτικοί. Είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανοχή 0% για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στις ζωοτροφές. Κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην αγορά. Ε, τα απλή που μεταφέρουν τέτοιε ουσίε αγκάζονται και επιστρέφουν πίσω, κάτι το οποίο σημαίνει 200 εκατομμύρια ευρώ απώλεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολλοί αρνούνται γενικά να μεταφέρουν σόγια γιατί φοβούνται ότι θα αναγκαστούν να γυρίσουν πίσω και τι θα γίνει, πώς θα αντικατασταθούν ε, αυτές ε, οι ζωοτροφές. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια συνέπεια που κάθε άλλο παρά είναι και οφείλεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πρέπει να αλλάξει λοιπόν αυτή η νομοθεσία για την μηδέν ανοχή και να, επιτραπεί η επιτραπούν οι ζωοτροφές αυτές. Σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε εργασίες επιτροπή πείς μας ραντεβού Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι. υπενθυμίζω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα είναι 9-10 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ όλους και τα λέμε στο επανειδήν.